Hello. Καλησπέρα σας και πάλι, συνάδελφοι. Καθίστε παρακαλώ και ετοιμάστε τις κάρτες ψηφοφορίας σας για να ξεκινήσουμε την απογευματινή μας συνεδρίαση. Είστε έτοιμοι? Φαντάζομαι προς... πως ναι. Θα ψηφίσουμε πρώτα την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους επίμονους οργανικούς ρήπους. Αναδιατύπωση και απόφαση. Τροπολογία 2. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 28. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 31. Υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται τροπολογία 3 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται ψηφοφορία. Γιατί είναι διαφορετικό σχετισμός δυνάμεων από το πρωί. Πρέπει να το ελέγξω κάποια δύο ψηφοφορίε. Είναι πολύ ωριακό το αποτέλεσμα. Απορρίπτεται πάντω. Τροπολογία 32. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 33. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 40 και 41 ποιος είναι υπέρ κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος για τις τροπολογίες 40 και 41, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας, εγκρίνονται. Τροπολογία 6, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές. Οι φιλελεύθεροι δεν ψήφισαν. Υπέρ εγκρίνεται. Τροπολογία 42 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 44 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 46 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 47. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τι 46. Οι σοσιαλιστές και το έλκυ ήταν κατά. Δεν κοιτάξατε.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 που σας τη μοιράσαμε. Είναι κανείς κατά. Έχουμε 5, 6, 7, 8 ενστάσεις κατά τις προφορικές τροπολογίες, οπότε δεν μπορούμε να την ψηφίσουμε. Ψηφίζουμε λοιπόν την 7 χωρίς την προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 55 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ Θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο για την 13. Πολύ ευχαρίστω. Γιατί έχω και εγώ κουραστεί και δεν είμαι σίγουρη για το αποτέλεσμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Α, το ΕΛ και οι σοσιαλιστές ψήφισαν κατά όντως, οπότε απορρίπτεται. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 14. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16 και 17 μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τροπολογία 18. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Μόνο την ένα την ψηφίσαμε, τη συμβαστική. Τροπολογία 19. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 21 υπέρ. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 20. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 24. Υπέρ. Κατά. Εποχές απορρίπτεται. Και τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. τη ψηφοφορία. Τέλος, εγκρίνεται. Περνάμε στο επόμενο θέμα. ψηφίζουμε την οδηγία με θέμα την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών. Ξεκινάμε με τη συμβαστική τροπολογία 2. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 150 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 151 και 152 και 127 ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται. 154 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τραν 28 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ποιο είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορία Και απορρίπτεται. 155. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 156 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 157 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 158 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τραν 29 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα. Τέλος. Και απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 8. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 166. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 167. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 167. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 168 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 169 και 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Περνάμε στη σελίδα 12 κατευθείαν. Έτσι μου λέει η γραμματεία. Συμβαστική τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τραν 40 υπέρ. Τραν 40 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 23 και 233. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 236 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 241 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 241 άρχεται η ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας απορρίπτεται Τραν 41 και 242. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. 244 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 251 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 245 και 249 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 250. Καταπίπτει. 246 υπέρ. Κατά. εποχές Απορρίπτεται. Τραν 43 υπέρ. Κατά. εποχές Εγκρίνεται. 252 252. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στη σελίδα 18. Και στην τροπολογία 280. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 281 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Τραν 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο για την 281. Πολύ ευχαρίστως. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Αυτό δεν είπα. Βοηθήστε με κι εσείς, γιατί όλοι ψήφισαν εκτός από τους συντηρητικού μεταρρυθμιστές. Λες και το έκαναν επίτηδες. Εν πάση περιπτώσει, ίσως εγώ βιάζομαι και δεν προλαβαίνετε να σηκώσετε τα χέρια. Τραν 49, ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τραν 50, ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 286 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 287 και 288. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τις ε, τροπολογίες 287 και 288. Άρχεται ψηφοφορία. Γιατί ψηφίζετε αλλιώ τώρα. Σκόπιμα το κάνετε. Ήβο. Γιατί ψηφίσατε έτσι. Επίτηδες. Τέλος, εγκρίνεται. Μα για την ομάδα η σύσταση ήταν ε, αρνητική ψήφος. Βλέπω, ο ένας κοιτάζει τον άλλον. Εγκρίνεται πάντως. Κύριε Λίζα, Δείξτε στην ομάδα σας πώς θα ψηφίζει. Με μπερδεύετε όταν υπάρχουν αντιφατικά μηνύματα. Συμβαστική τροπολογία 6. Ποιος είναι υπέρ. Υπέρ για τη συμβαστική 6 κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη συμβαστική τροπολογία 7. Τέλος. Απορρίπτεται όντως. Συμβαστική τροπολογία 5. εμείς Συμβαστική 5, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη συμβαστική τροπολογία 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Εδώ είναι άλλη ισορροπία δυνάμεων. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται ισοπαλία. άρα θα έχουμε άλλες τροπολο... πολλές τροπολογίες να ψηφίσουμε. Πόσες. Σωστά ψήφισε αυτή τη φορά. 291. Τώρα πρέπει να ψηφίσουμε τις επιμέρους ε, τροπολογίες. 291. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 292. 289, συγγνώμη. 289. Η συμβαστική τροπολογία 5 απορρίφθηκε. Ναι, αλλά η 6 εγκρίθηκε. Α, δίκιο έχετε. Μπράβο, Ρενάτε. Οπότε, Πηδάμε στη σελίδα 26. Από ό,τι φαίνεται, εκτός και αν έχετε αντίρρηση. Τροπολογίες 34 και 35. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τραν 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 37 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 37 38 και 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 40 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τραν 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τραν 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τραν 4. Τμήμα 1 υπέρ. Κατά αποχές. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία and it is closed. Oh, it was adopted. 40... Εγκρίνεται. Ε, η 42 καταπίπτη. Τραν 4, τμήμα 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 47. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 51 και 52 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 36 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τραν 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν βλέπω την κουέ. Τραν 7. Υπέρ. Εγκρίνεται. Τραν 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 56. Και τραν 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 57. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τραν 9, τμήμα 1. Υπέρ. Όχι. Καταπίπτει. Τραν 9, ε, τμήμα 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 59. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 60. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τραν 12 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 64 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τραν 13 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 69. Θέλετε να ελέγξουμε την 67 ηλεκτρονικά. Ωραία. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας. Τυχερή ήμουν τελικά. Όντως απορρίπτεται. Αλλά πρέπει να πω ότι την ΚΟΕ δεν την είδα. Πρέπει να σηκώνετε τα χέρια σας λίγο πιο ψηλά μάλλον. 69. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία. 1 και 72. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 73. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Καταπίπτει. Α, α, είναι ταυτόσημη. Συγγνώμη, ήταν στην άλλη σελίδα. Ε, 74. Απορρίφθηκε νομίζω. Λοιπόν, 74. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Πέρα της προφορίας. Εγκρίνεται. Μετά πάμε στην 78 τμήμα 1 υπέρ. 78, τμήμα 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τμήμα 2. Υπέρ. Α, καταπίπτει. 79, τμήμα 1. Καταπίπτει. Δεν καταπίπτει. 79, τμήμα 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. It's a cross close. It is adopted. εγκρίνεται. 79 τμήμα 2. Υπέρ, κατά, αποχές. Δεν μπορώ να πω. Το ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας Πέρας ψηφορία. Απορρίπτεται. Some didn't vote, huh? just for your information. Because we see the... Κάποιος δεν ψήφισε. 3. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Α, συγγνώμη, καταπίπτει 3. Πάμε στην 4 και 92. Ταυτόσιμες. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Τραν 16. Υπέρ, κατά, αποχές, να το ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ναι, αλλά άλλοι έχετε καταψηφίσει. Το ξέρετε, έτσι. Τραν 16. Την Τραν 16 ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορία και εγκρίνεται. Αλλά πραγματικά νομίζω ότι σηκώσατε στο κατά τα χέρια σας. Τέλος πάντων. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 90, όχι, τραν 11, υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Τραν 10, υπέρ. Κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 90, όχι, καταπέπτει 96. Τραν 17, υπέρ. Κατά, αποχές απορρίπτεται. εκατό, υπέρ, κατά, αποχές, να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. We, we vote on this 102 and 5. Uh, it's closed. Πέρας ψηφοφορίας. Βλέπετε τι γίνεται, απορρίπτεται. Η τρίτη με το ίδιο αποτέλεσμα. Δεν καλύπτονται από το πέντε, οι επόμενες. Εκατόν τέσσερα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ενενήντα 99. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 105 υπέρ κατά ελέγχουμε την 105. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τράνα 18 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 106 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 109 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε την 109. And it is uh, closed. εγκρίνεται. Τραν 19 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τραν 20 υπέρ, καταπίπτει, δεν εγκρίθηκε 29. Τραν 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 115 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 116 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 118 και 119 ταυτόσημες υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 122 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 123 και 128 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 125 Η 10 εγκρίθηκε. Άρα καταπίπτει 125. 126 και 127. ταυτόσιμες υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 129 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 131 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 132 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 325 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 136 και τραν 24 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 141 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τραν 23 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 148 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 100... Α, 148. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 148. Άρχιτη ψηφοφορία. Ναι, αλλά οι πράσινοι υπερψηφίσατε. Πέρας ψηφοφορίας εξεκολουθεί να εγκρίνεται. 149 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τραν 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τελική ψηφοφορία για το σύνολο της έκθεσης. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Και πέρας και εγκρίνεται. That was a difficult one. Yeah, yeah. that's why I didn't want to put it together with plastics in the morning. <laughs> Bună, Ștefan. Okay, now we vote on... Uh... Πότε ψηφίζουμε για την επόμενη έκθεση ευθυγράμμιση των ε, υποχρεώσεων αναφορών στα θέματα περιβάλλοντος. Τροπολογία Άγκρι 6. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος. The vote Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 8. Και άγκρι 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Εννέα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος. Έναρξη. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Γιούρι 4. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Γιούρι 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγ, απορρίπτεται. Άγκρι 8 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 43 και Γιούρι 7 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Γιούρι 8 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άγκρι 13 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Γιούρι 12 υπέρ, κατά, αποχές, το... οι σοσιαλιστές δεν έδειξαν, δεν ψήφισαν. Γιούρι 12 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 53 και Γιούρι 16, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 55 υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος για την 55 έναρξη ψηφοφορίας και πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άγκρι 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Γιούρι 19 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 60 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 61 και άγκρι 15 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Γιούρι 22 υπέρ κατά, αποχές, έλεγχος. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Γιούρι 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Γιούρι 24 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 68 και άγκρι 16 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 69 και άγκρι 17 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Γιούρι 25 υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται, Γιούρι 26 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 70 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 27 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, Οπότε περνάμε στην 22 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Γιούρι 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 71. Έχουμε προφορική τροπολογία από την ομάδα των Πρασίνων. Είναι κανείς ε, που αντιτίθεται, έχει αντίρρηση. Όχι, από ό,τι ψηφίζουμε ε, για την 71 μαζί με την προφορική υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Γιούρι 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Γιούρι 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 23 και 73 και Γιούρι 31 υπέρ κατά αποχές απορι, εγκρίνεται. 74 και Γιούρι 32 υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Και εγκρίνεται. Άγκρι 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άγκρι 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Πέρας ψηφοφορίας. Και εγκρίνεται. Γιούρι 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 24 υπέρ. Κατά. Έλεγχος για την 24. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Γιούρι 34 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Γιούρι 35 υπέρ. Κατά αποχές δεν ξέρω έλεγχος. Πέρας. Εγκρίνεται. 36. Ποιος είναι υπέρ? Την, ψηφί... Την ψηφίσαμε 35, 36 τώρα, 36. Κατά, αποχές απορρίπτεται. 77 και άγκρι 21. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 25 και 76. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στη Γιούρι 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Γιούρι 38. Τι κάνουμε. Γιούρι 38. Πρέπει εγώ να σας πω, ε. Ναι. Ως εισηγήτρια. Πέρας ψηφοφορίας και εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 27 και άγκρι 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. άλτε, Υπέρ. Εγκρίνεται. Η 79 και Γιούρι 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ογδόντα και Γιούρι 41 ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Γιούρι Σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος της Γιούρι 1, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 30 και άγκρι 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 38 και γιούρι 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Άγκρι 5 υπέρ κατά Αποχές. Εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται ηλεκτρονικά για την τελική ψηφοφορία έναρξη. Πέρας. Και εγκρίνεται... is different. <laughs> okay. Um, now we are voting on the resolution for COP24. Περνάμε τώρα στο ψήφισμα για την COP24, τροπολογία 20. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 26, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 3, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 33, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας και εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 46. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 57. Περ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 60 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Άρχεται η ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Δύο ομάδες τουλάχιστον ήταν κατά. Ήταν τεράστια διαφορά.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 Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 66 έξι υπέρ. 66 λέω υπέρ κανείς ούτε ένας κατά αποχές απορρίπτεται 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 87 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 89 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 95 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 100 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 101 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 101 άρχεται ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 104 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 105 κατά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 110 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 110 άρχιτη ψηφοφορία Έγκρινεται. 111 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 113 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 114 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 115 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και αυτό 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 117 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 118 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 120 120. Ποιος είναι υπέρ? Κατά αποχές εγκρίνεται. 121 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 122 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 123. Ποιος είναι υπέρ? Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 10. Ποιος είναι υπέρ? Κατά αποχές εγκρίνεται. 125 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 126. Ποιος είναι υπέρ? κατά αποχές απορρίπτεται. 128 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 129 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 130 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 131 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 132 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 133 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 134 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 135 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 136 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα έχουμε τις τροπολογίες της ΔΕΒΕ. Θα λέω την παράγραφο. Για την παράγραφο 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 5. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος. Τέλος ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Παράγραφος 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 8. Υπέρ. Κατά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 κατά αποχές εγκρίνεται. Δύο υπέρ κατά αποχές δεν ξέρω Ελεκτρονικός έλεγχος για τη δύο. άρχεται η ψηφοφορία τέλος εγκρίνεται τροπολογία τρία. ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 σε 2 τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ,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 απορρίπτεται 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Δεύε για την ιδεολογική σκέψη 1 ποιος είναι α ποιος είναι υπέρ κατά το έλκτη είναι υπέρ ή κατά τότε εγκρίνεται αφού είστε υπέρ Φαντάζεστε, μετράει η ψήφο σα. Για το β, β αιτιολογική σκέψη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σ α, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δ α, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Φ. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. I υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. J υπέρ κατά Υπάρχουν και ψήφοι κατά του J. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την αιτιολογική σκέψη J. εγκρίνεται και τελική ψηφοφορία για το ψήφισμά μας ηλεκτρονικά. Παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και άλλες ψηφοφορίες έχουμε. Πέντε ακόμη. Παρακαλώ, ζητώ τη συνεργασία σας. Έχουμε πολλές ψηφοφορίες σήμερα. Okay, so first we vote. Λοιπόν, πρώτον θα ψηφίσουμε για τον κανονισμό για το πρόγραμμα πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας που θεσπίζει τους κανόνες συμμετοχής και διάδοσης είναι συναπόφαση. Ξεκινάμε από την, 10, από την 78 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 79 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 80 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 82 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 105 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 106 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 107 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 108 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 109 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 110 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 111 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 112 έχει προφορική τροπολογία των πρασίνων. Αντιτίθεται κανείς την προφορική. Αν όχι, ψηφίζουμε μαζί με την προφορική 112 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 205. Το ίδιο. προφορική τροπολογία. Αντιτίθεται κάποιος. Όχι. Ψήφος από κοινού. 205 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 9 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 119 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 120 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 12 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Σελίδα 11 τώρα. Συμβιβαστική 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Σελίδα 13, 183, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 15, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 16, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 184, υπέρ, κατά, Αποχές απορρίπτεται. 185 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 186 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 187 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 188 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 189 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 190 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 191 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 192 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Έναρξη. Και πέρας. Εγκρίνεται. 193 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 194 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 195 υπέρ. Κατά αποχές δεν είναι σαφές. Έλεγχος. 195. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 196 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 197 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 198 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 199 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 200 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 201 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 203 υπέρ, κατά, έλεγχος. Πέρας. Εγκρίνεται. 204 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 207 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 212 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.13 και 2.14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2.15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2.17 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.19 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.20 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 2.21 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 26 υπέρ, κατά, α, έλεγχος. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. 2.23 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος για την 27. Πέρες. Απορρίπτεται. 2,25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2,26 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 227 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 228 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 230 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 231 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 234 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.35 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Έναρξη και πέρα ψηφοφορίας και εγκρίνεται. 2.36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.40 και, 28. 2.40 και 28 μαζί υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 29 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2.42 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2.43 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2.44 υπέρ. Κατά έλεγχος. Για 2.44 πέρας εγκρίνεται. 2.45 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά αποχές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 κατά, αποχές, εγκρίνεται. 4. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 47 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 51 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 52 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 54 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 55 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 56 υπέρ, κατά, απο... το ΕΛΚ τι είναι, υπέρ, τότε εγκρίνεται. 57 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 58 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 61 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ κατά. Κανείς. 62 υπέρ Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 70 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 75 υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος για την 75. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά έναρξη. Και πέρας. Και εγκρίνεται. Τώρα θα ε, ψηφίσουμε επί της απόφασης για τη δημιουργία... Α, το συγκεκριμένο πρόγραμμα της ε, υλοποίησης του Horizon Europe. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Σελίδα 4. Συμβαστική 3. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά, τροπολογία 88, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 89 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 90 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 92 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 95 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 99 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 100 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 101 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 102 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχέ. εγκρίνεται. Έχουμε προφορική τροπολογία στην 107. Έχει κάποιο αντίρρηση. Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν από κοινού με την ε, προφορική. Τροπολογία 107. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 108. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 109 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 110 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 111 όχι πίπτη. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 112 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 12. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 6. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 115. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 116. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 117. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 119 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 118 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 120 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 121 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 122 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 123 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 124 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 125 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 126 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 128 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 135 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 136 υπέρ κατά καταπίπτει. Καταπίπτει. Μετά πάμε στην 18. Τροπολογία 18 στην επόμενη σελίδα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 139 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 144 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 145 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 146 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 157 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 158 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Την 158. με κοροϊδέψατε. Ε, Ε, 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 161. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 163 και 164 ταυτόσημες υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 165 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 166 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 167 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 168 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 169 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 170 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 172 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 173 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 174 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 175 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 176 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 177 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 178 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 179 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 33 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 180 υπέρ κατά. Το ΕΛΚ άρα εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 181 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 39 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 186 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 187 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 188 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 189 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 190 ε, υπέρ κατά αποχές απο, α, ε, α, απορρίπτεται. 191 υπέρ κατά εγκρίνεται. 192 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 193 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 194 υπέρ κατά να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ. 195 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 196 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 197 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε τις 42 ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται. 198 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ κατά αποχές Άλτε. υπέρ εγκρίνεται. 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 201 και 202 και 203 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 204 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 205 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 45 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 206 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 207 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 208 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 46 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 209 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 210 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 47 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 211 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 212 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 213 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 214 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 215 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 216 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 217 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 218 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 219 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 220 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 221 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 222 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 223 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 224 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 227 υπέρ. Κατά αποχές. Δεν ξέρω. Υπέρ. 227 υπέρ. Εγκρίνεται λοιπόν. 228 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 229 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 230 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 231 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 232 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 56 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 57 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 58 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 60, 59, συγγνώμη, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 60 ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 61 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 63 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Και ψηφίζουμε τελη... τε... τελική ψηφοφορία για το σύνολο της έκθεσης. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας και εγκρίνεται. I appreciate the part with the compromises very much. Um, Ψηφίζουμε επί της απόφασης του Συμβουλίου για την σύναψη σχέση, Εταιρική συμφωνίας Ευρωπαϊκή σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, η τροπολογία είναι ποιο είναι υπέρ. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Έναρξη τη ψηφοφορία. Τροπολογία 1. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Σχέδιο γνωμοδότησης όπως τροποποιήθηκε έναρξη ψηφοφορίας. Ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται.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 απορρίπτεται. 22 υπέρ κατά απορρίπτεται. 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε για, για το τελικό κείμενο ηλεκτρονικά. Έναρξη και πέρας. Απορρίπτεται.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 Απορρίπτεται. Και τώρα η κυρία Μελά έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αυτή η φοβερή λιτανία απορρίψη, απορρίπτεται, απορρίπτεται, είναι εφαρμογή της δημοκρατίας. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κρίμα που στην έκθεση αυτή, που ήταν αξιολόγηση της υλοποίησης, έχουν γίνει διάφορες εκδόσεις. Τρεις εκθέσεις της Κομισιόν είπαν ότι το αποτέλεσμα δεν ήταν ε, το αναμενόμενο ακριβώς και κυρίως λόγω του βάρους του τίτλου 9 του εμπορίου και της βιώσιμης ανάπτυξης σε μια στιγμή που οι χώρες της Νότιας Αμερικής βρίσκονται σε φάση ε, πιθανής ε, οικονομικής αποσταθεροποίησης δεν μπορούμε να, δώσουμε, να γνωμοδοτήσουμε για την Κομισιόν επί της ουσίας. Φυσικά το θέμα δεν είναι πάντα ε, δεν έχει σχέση με την πολιτική. Δεν νομίζω ότι αυτού του είδους συμπεριφορά είναι η τρίτη έκθεση σε λιγότερο από μία εβδομάδα που αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο, ότι αυτό ενισχύει την δημοκρατία και επιτρέπει κάποιους να βρίσκονται εδώ, θα επιτρέψει σε κάποιους να βρίσκονται και πάλι εδώ τον Ιούλιο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ολοκληρώνεται οι ψηφοφορίες καθώς και η σημερινή συνεδρίαση. Αύριο το πρωί στις 9. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.